την έκθεση Καριμά Ντελή σχετικά με την αστική κινητικότητα. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγο καιρό το 80% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ζουν σε αστικές περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν η μετακίνηση των ανθρώπων αυτών να διευκολύνεται για αυτούς που πηγαίνουν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να αναζητήσουν εργασία, να πάνε στο γιατρό τους, στον οδοντίατρό τους, στον κινηματογράφο ή στο αθλητικό γήπεδο. Υπάρχει λοιπόν ένα δικαίωμα στην κινητικότητα, αλλά θα πρέπει η κινητικότητα δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο επιλογής αλλά είναι κάτι το οποίο θα έλεγα επιβάλλεται λόγω της καθυστέρησης, λόγω της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Οι πόλεις θα έλεγα δημιουργήθηκαν τελικά για τα αυτοκίνητα και όχι για τους κατοίκους τους. Υπάρχει κλιματολογικό πρόβλημα, σας θυμίζω την COP21. Στις Βρυξέλλες ε, οι μαζικές μεταφορές είναι 25% ε, του συνόλου των εκπομπών. Λοιπόν, θα πρέπει ε, να υπάρξει αλλαγή σε σχέση με τους στόχους μας μέχρι το 2030. Το 2015 το να αναπνέει κανείς σκοτώνει. Χιλιάδες θάνατοι κατέτος από ε, τα σωματίδια των πετρελαιομηχανών. Ε, φύγουν και σκοτώνουν τα παιδιά της ε, γυναίκες, τους ηλικιωμένου και φύγουν φυσικά τους πνεύμονες τους και ο θάνατος από τη μόλυνση την αναπνευστική είναι κύρια αιτία θα έλεγα για την απώλεια ανθρώπινης ζωής στον 21ο αιώνα και θα σταματήσουμε τα πράγματα να εξαρτώμεθα και από τις πετρελαϊκές δικτατορίες. Ε, ταυτόχρονα ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα ε, συμβαίνει σε αστική ε, περιοχή και υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. 25 εκατομμύρια νοικοκυριών έχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με την κινητικότητα, δεν έχουν πρόσβαση σε μαζική μεταφορά ή είναι δύσκολη η πρόσβαση αυτή γιατί μπορεί να είναι πάρα πολύ ακριβή. Είναι λοιπόν εφικτή μια νέα κινητικότητα. Δεν είναι μόνο εφικτή, είναι απαραίτητη. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ε, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές και δημοκρατικές επιπτώσεις των μεταφορών και για μας αλλά και για τις επόμενες γενιές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει φιλόδοξους στόχους και στα πλαίσια λοιπόν της COP21 θα πρέπει η ε, αποδοτικότητα η ενεργειακή να οδηγήσει στην ε, απαγόρευση χρήσης του πετρελαίου ε, και το 2050 της ε, κατάργησης των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων. Να υπάρξουν ε, μέσα μεταφοράς ηλεκτρικά όπως τραμ, τρόλεϊ, να περάσουμε από τον δρόμο στον σιδηρόδρομο, να περάσουμε από τον δρόμο ακόμα και στις παραποτάμιες συγκοινωνίες, να περάσουμε στις πολυτροπικές συγκοινωνίες Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μπροστά μας, υπάρχουν τεράστια λόμπι. Υπάρχει το αυτοκινητιστικό λόμπι που είναι υπέρ του status quo και δεν θέλουν να ανοίξει τίποτα και να αλλάξει τίποτα. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για μια φιλόδοξη νομοθετική πρόταση αν θέλουμε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δική σας Επιτροπή να είναι η Επιτροπή της τελευταίας ευκαιρίας όπως λέει ο Πρόεδρος Γιούνκερ. Οι Ευρωπαίοι εμάς περιμένουν, πρέπει να προχωρήσουμε και ας μην τους απογοητεύσουμε γιατί αλλιώς η κινητικότητα σε αστικές περιοχές είναι ένα βασικό πρόβλημα και πρέπει να χαρακτηριστεί σαν βασική προτεραιότητα. Η κυρία ε, Μπούλτση, η Επίτροπος Μπούλτση έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Αξιότιμε, αξιότιμες και αξιότιμοι ευρωβουλευτές έκθεση που θα εγκρίνεται σήμερα αποτελεί προϊόν καρποφόρου εργασίας. Είναι συνεκτική, εμπνέει και σε μεγάλο βαθμό ευθυγραμμίζεται σημαντικά με την ε, νοοτροπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ όλα τα πρόσωπα που συνεργάστηκαν για την έκθεση και 500 τροπολογίες που κατατέθηκαν δείχνουν πόση προσπάθεια, πόσο κόπος απαιτήθηκε για να εκπονηθεί η έκθεση. Έκθεση που δείχνει ότι τα αστικά κέντρα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία για όλες και όλους μας. Πολύ απλά διότι όλο και περισσότεροι από μας ζούμε σε αστικά κέντρα, πάνω από 80% των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα είναι λογικό να αντιμετωπίζουμε και σημαντικές προκλήσεις. Σημαντική αριθμή προσώπων, δυσκολίες στην ε, κίνηση, στην κυκλοφορία, διοξιδία του άνθρακος κλπ. Όλα αυτά τα απηχεί εκθεσή σας και προτείνει μάλιστα και λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν. Δεν θα τις συζητήσω όλες αυτές. Έρχομαι μόνο σε τρεις που μου φαίνονται πολύ σημαντικές. Πρώτα, η βιωσιμότητα των αστικών συγκοινωνιών που αποδείχτηκαν πολύ σημαντικές εθελοντικά μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν. Αυτό ενθαρρύνει, μας ενθαρρύνει στις προσπάθειές μας στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ε, υποβολή μάλλον ε, κατευθυντήριων γραμμών. Προσπαθήστε και επιτόπου. Εφή συστήματα μεταφορών. Δεύτερος τομέα. Ίσως να γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μία πλατφόρμα για ιδέες που να εφαρμοστούν όσο γίνεται γρηγορότερα. Τα αστικά κέντρα θα ωφεληθούν πολύ και γενικότερα η έκθεσή σας αναγνωρίζει και το τεράστιο δυναμικό που προσφέρει η ψηφιοποίηση για τα συστήματα μεταφορών και συγκοινωνιών. Η ψηφιοποίηση των μεταφορών είναι προσωπική κιόλα προτεραιότητα δική μου. Ο τρίτος τομέας, δηλαδή επενδύσεις και καινοτομία, που και τα δύο αυτά επιτρέπουν και τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης. Πώς θα προσελκύσουν περισσότερες επενδύσεις στα αστικά κέντρα, πώς θα αυξήσουν την καινοτομία, πώς η καινοτομία θα στηρίξει την βιωσιμότητα. Η έκθεσή σας επιβεβαιώνει ότι η καινοτομία στις αστικές συγκοινωνίες προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες. Ας σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η μείωση των διοξιδιών του άνθρακου σημαίνει υψηλά κόστη. Με την αστικοποίηση που είναι η παγκόσμια τάση Είμαι πεπισμένη ότι όλες αυτές οι προσπάθειες θα αποδώσουν και θα συμβάλλουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Ανάπτυξη και Νέες Δουλειές. Τώρα για το FC, που είναι μηχανισμός για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αστική ε, κινητικότητα είναι πλουσιότατο θέμα. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολύ περισσότερα πράγματα. Ασφάλεια, τροχιά ασφάλεια δηλαδή, η ΣΕΦ, άλλα ε, ε, ταμεία συνοχής και ούτω καθεξής. Όμως, τώρα έχει έρθει η ώρα να συζητήσετε εσείς. Αναμένω λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις και τα σχόλιά σας και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω στη, στο τέλος της συζητήσεώς σας σε ό,τι θέλετε να μου θέσετε υπόψη. Η Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, θα πρέπει να επενδύσουν οι πόλεις ε, για να αποφύγουμε την ε, συμφόρηση. Είναι σημαντικό για την οικονομία, για το περιβάλλον και για μας τους ίδιους τους πολίτες. Ε. Αποτελεσματική κυκλοφορία. Αυτό χρειαζόμαστε για την εξοικονόμηση κιόλας των δαπανών για την αντιμετώπιση της μόλυνσης. Ε, πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα μεταφοράς, όχι μόνο το αυτοκίνητο, αλλά και ποιότερους τρόπους μεταφοράς, ε, όπως το τραμ, τα ποδήλατα, τα λεωφορεία, τα τρένα. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις και για το ΕΛΚΑ είναι σημαντικό οι πολίτες να προκρίνουν τις λύσεις που είναι φιλικότερε προς το περιβάλλον. Χαιρόμαστε που ακούμε αυτές τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Εξάλλου η ψηφιοποίηση προσφέρει και νέες δυνατότητες για την ε, κοινή μεταφορά, την ευφυή e e μεταφορά, για το Uber Share, Χρειαζόμαστε νέες λύσεις ε, χάρη στι νέε τεχνολογίες που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Άντερσον, μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη όλη την ποικιλομορφία των αστικών, περιαστικών και υπεθρίων ζωνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υποβάλλει τις νέες προτάσεις της. Υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα μεταφοράς ε, και διαφέρουν ε, ανάλογα με την περιοχή όπου κατοικούν οι πολίτες μας. Εγώ χαίρομαι διότι με την έκθεση ασχολούμαστε με το θέμα των μεταφορών εμπορευμάτων. Ε, οι αστικές ζώνες αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα των εκπομπών. Σωστά το είπατε και άρα χρειαζόμαστε κινητικότητα και για μα και για τι μεταφορέ και για την οικονομία μα. και θα ήθελα τα σχόλιά σα γι' αυτό επίση. ζητάτε ε, για την διαχείριση της η κυκλοφορία και για τα μέτρα εφαρμογή. Πολύ θετικό καλωσορίζουμε αυτό το μέτρο. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι συνιστά πρόβλημα οι ασφαλές οδικές μεταφορές. Πολλοί πολίτε και ποδηλάτε Τραυματίζονται ή σκοτώνονται στι πόλει μα στην Ευρώπη κάθε μέρα. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Επίση, στι πόλει βλέπουμε μεγάλα χάσματα ανάμεσα στου έχοντε και του μη έχοντε. Χρειαζόμαστε καλέ δημόσιε μεταφορέ. Αυτό έχει σημαντικά οικονομικά και οικονομικά ε, ωφέλη και ε, για την πρόσβαση επίση στην αγορά εργασία και για να εξέρχονται από την παγίδα τη φτώχεια οι πολίτε. Υπάρχουν πολλέ μακροπρόθεσμε προτεραιότητε από πλευρά μα και τι λαμβάνει εν μέρη υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μόνο μία τροπολογία σε αυτή την έκθεση και καλούν του συναδέλφου να την εγκρίνουν. Συμφωνούμε όλοι για το phasing out, σταδιακή κατάργηση των σημαντικών καυσίων. Παρακαλώ να ε, υπερψηφίσετε την τροπολογία. Τώρα, από την πλευρά των συντηρητικών, ο κύριο Τονεσόφσκι. Ευχαριστώ. Επίτροπε, είμαι πρώην δήμαρχος μιας μεγάλης πόλης και πρώην περιφερειάρχης στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Έχω μεγάλη εμπειρία στον τομέα της αστικής κινητικότητας και έχω έρθει σε επαφή με πάρα πολλούς φορείς σε πολλά μέρη της Ευρώπης και ξέρω πως ε, υπάρχουν ε, ε, ιστορικά σημεία αναφοράς και ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν σε κάθε περιοχή. Ευχαριστώ την Επιτροπή την εισηγήτρια για την έκθεσή της και την ευχαριστώ επειδή συμπεριέλαβε κάποια από τα σχόλιά μας. Ε, παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να έχω κάποιες αμφιβολίες ε, σε σχέση με την ευφυή αστική κινητικότητα ως προς τους πετρελοκινητήρες ε, αλλά και τους βενζινοκινητήρες. Πρέπει να υποστηρίξουμε την αστική κινητικότητα με άλλους τρόπους. Σας ευχαριστούμε. Έχετε γαλάζια κάρτα, τη δέχεστε, ωραία. Αγαπητέ συνάδελφε, εάν κατάλαβα καλά, από ό,τι κατάλαβα συμφωνείτε με τα μέτρα κατά των πετρελαιοκινητήρων. Είσαστε υπέρ όμως της αστικής κινητικότητας. Πώς ακριβώς το εννοείτε. Προτείνετε συγκεκριμένα μέτρα, κύριε Τονασεύσκη. Μικρό,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 Σίγουρα ε, με τα μέτρα βιωσιμότητας της αστικής κινητικότητας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η αστική κινητικότητα. Όμως ε, το να καταργήσουμε δια μιας συγκεκριμένους τύπους κινητήρων δεν είναι η λύση. Η απεξάρτηση από τον άνθρακα μπορεί να ακολουθήσει εναλλακτικέ οδούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε δύο-τρία χρόνια στην αυτοκινητοβιομηχανία. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί και ταπεινοί κυρίως ως προς την επιστημονική πρόοδο που μπορεί να επιτευχθεί τα επόμενα δύο-τρία χρόνια. Ευχαριστούμε. Βαν Ευχαριστώ. Κάθε ευρωπαϊκή πόλη είναι και διαφορετική. Βεβαίως, ζητήματα κινητικότητας έχουν όλες. Βεβαίως η Ευρώπη πρέπει να δώσει στόχους και αν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς που πρέπει να είναι η ασφάλεια των ε, τροχιών μεταφορών, βεβαίως πρέπει να ε, βρούμε και ευφυή συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ των τα αυτοκίνητα, να, είναι, ε, υπάρχουν τραμ και άλλες καθαρές μεταφορές, αλλά όλα μπορούν να γίνουν και φθηνότερα και ευφιέστερα. Να πάρουν το ποδήλατο οι Ευρωπαίοι μέσα στα αστικά κέντρα. Οι αποστάσεις είναι μικρέ συνήθως. Καλύτερα λοιπόν να παίρνουν το ποδήλατο παρά το αυτοκίνητό τους. Καλύτερα και για την υγεία τους και για το πορτοφόλι τους. Και βεβαίως εν τέλει και για το περιβάλλον. Αυτά οφείλετε να τα γνωρίζετε. Αυτό θα σημάνει πραγματική βιώσιμη κινητικότητα. Ο επόμενος συνάδελφος για ένα λεπτό. Κυρία Κίλονεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων προκαλεί και το 25% του διοξιδίου του άνθρακος και βεβαίως και πολλά άλλα προβλήματα, πολλές άλλες επιβλαβείς ουσίες. Εδώ πρέπει να κάνουμε σοβαρή προσπάθεια. Ωστόσο, ωστόσο είναι λυπηρό που δεν υπάρχει δηλωμένη θέληση από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν. Η επικουρικότητα βεβαίως είναι σημαντική αρχή. Πολύ συχνά όμως πίσω από την επικουρικότητα κρύβεται μόνο μια αδράνεια των χωρών μελών που δεν επιθυμούν να αλλάξουν τα κακό σκήμενα. Βασική πηγή των ε, ρήπων ε, στα αστικά κέντρα είναι το αυτοκίνητο. Και αυτό που προσπαθούν ορισμένοι να κάνουν εδώ είναι να το υπερασπιστούν κι άλλο. Το αυτοκίνητο όμως απειλεί την ποιότητα ζωής στις ε, πόλεις μας. Χρειάζεται να, βρει, να βρεθεί κάποια λύση. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι διατεθειμένη να λάβει δραστικά μέτρα. Βόιτ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στην αιτιολόγηση του ψηφίσματος λέγεται ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση στις χώρες μέλη να μεταφέρουν την κίνηση από την τροχιά κυκλοφορία στο σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει όμως κανένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Πολλές πόλεις μπορεί κανείς σε, να κυκλοφορήσει, να φτάσει μέχρι αυτές δηλαδή και από υδάτινες οδούς. Αυτό θα ήταν προτιμητέο. Τώρα και για το σιδηρόδρομο εγώ βλέπω το αντίθετο. Εδώ και δύο χρόνια χιλιάδες λεωφορεία αναλαμβάνουν τις υπεραστικές συγκοινωνίες και οι επιβάτες εγκαταλείπουν τον σιδηρόδρομο και παίρνουν τα αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο σημαίνει έξτρα επιβάρυνση και για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και για το περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν περαιτέρω επεξεργασία της ε, ιδέας αυτής. Βάντε Κάμπ. Βάντε Κάμπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι κοινό μυστικό θα έλεγα ότι η διατήρηση η επεξεργασία και η διατύπωση της συγκεκριμένης πρότασης ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Και οι πράσινοι, σαν παράδειγμα, έχουν ξεκάθαρες απόψεις σε σχέση με την χωροταξία και την κινητικότητα σε αστικές περιοχές. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μία απάντηση απέναντι στα προβλήματα των πόλεων. Η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκαθαρίσει επίσης και τις αρμοδιότητες της σε σχέση με τον καθορισμό της συγκεκριμένης πολιτικής. Παρ' όλα αυτά οφείλουμε εμείς να καταστήσουμε τις πόλεις μας ομορφότερες, καθαρότερες ε, πόλεις τις οποίες να μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς αυτοκίνητα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια καλή πρώτη έκθεση. Ρεβόντα Λον Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η, κινητικότητα σε αστικές περιοχές συνδυάζει την οικολογία, την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Η κινητικότητα μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση ε, της, ε, ατμόσφαι, της μόλυνσης της ατμόσφαιρας. Βλέπουμε ότι η αστικοποίηση δυστυχώς συνεχίζεται και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε αιτήσια βάση και γι' αυτό θα πρέπει να καταστήσουμε την κινητικότητα αηφόρο. Ε, σε σχέση με την τροπολογία 1 που θέτει το θέμα των πετρελαιοκινητήρων, θα πρέπει να καταργηθούν οι ευνοϊκές για τους πετρελαιοκινητήρες ρυθμίσεις. Είναι ε, ε, απαραίτητο και λυπάμαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης ε, στην αρμόδια επιτροπή η κοινωνική διάσταση δεν ελήφθη όσο έπρεπε υπόψη. Ο κύριος Ζλοτόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, η ζωή στις πόλεις έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τα προβλήματα της μετακίνησης είναι γνωστά μποτιλιαρίσματα, ε, ατυχήματα αυτοκινητιστικά, ελλειπείς υποδομές μεταφορών. Είναι πράγματα που ε, σε καθημερινή βάση βιώνουν οι πολίτες. Όλα αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα εξαφανίσουμε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα μειώσουμε μέσω της χρήσης τραμ και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα καλύψουμε τις ανάγκες ε, των πολιτών και των πεζών φυσικά όπως και των ποδηλατών που θα πρέπει να την χάνουν υψηλότερης προστασίας. Είναι μια καλή πρόταση λοιπόν. Από την άλλη δεν συμφωνώ με κάποιες ε, θα έλεγα ε, στάσεις απέναντι στους οδηγούς των οχημάτων οι οποίες είναι θα έλεγα κακές. Κυρία Πρόεδρε, βεβαίως η αστική κινητικότητα είναι ζήτημα και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και κοινωτική στήριξη, Είναι όμως θέμα νομοθετικό για μα, μάλλον όχι. Γι' αυτό και προσπαθούμε να εξετάσουμε περισσότερο τα καυσαέρια κτλ. που πρέπει να συζητηθούν. Πάντω όχι σε τούτην εδώ την έκθεση. Και τα ποδήλατα, βεβαίω. Δεν έχουμε όμως ούτε και αρμοδιότητα. Και το Συμβούλιο Υπουργών για τις συγκοινωνίες δεν έχει τίποτα καλύτερες ιδέες παρά να στέλνει, το κόσμο, να τους υπουργούς με τα ποδήλατα. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες, ορισμένα ήταν και λογικά, τι μένει όμως απαγορεύσεις ε, κινητήρων ε, εσωτερικής καύσεως, απαγορεύσει κυκλοφορία σε κάποια Σαββατοκύριακα κτλ. Αντί για Κυριακές ελεύθερες από αυτοκίνητα, καλύτερα να ασχοληθούμε με τα προβλήματα των αστικών κέντρων και αντί για ποσοστώσεις ποδηλάτων, καλύτερα να ασχοληθούμε με ποσοστώσεις προσφύγων. Ευχαριστώ. Η κυρία Ταπαρντέλ, ένα λεπτό. Ε, υπάρχει θέμα στον τομέα των μεταφορών με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και τις επιπτώσεις που έχει και στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεψήφισε την πρότασή σας για τη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές και τώρα προτείνει και τις δικές του απόψεις για την αηφορία στην κινητικότητα των αστικών περιοχών. Εγώ για έξι χρόνια ήμουν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Βουκουρεστίου και νομίζω ότι στα πλαίσια της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης έχουμε την δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής καθιστώντας την κινητικότητα πιο αηφόρο και ταχύτερη. Μπορούμε να προτείνουμε λοιπόν μέτρα για πιο αποτελεσματική διαχείριση των μεταφορών ε, για τις συνοδευτικές επιμελητιακές υπηρεσίες και μέσω επίσης της σωστής κατάρτισης των πολιτών για εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Περνάμε στο Catch the Eye. Μοντέιρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πιστεύω πως πρέπει να προωθήσουμε την αστική κινητικότητα ε, με κίνητρα για την προώθηση των δημοσίων μεταφορών και προώθηση των μεταφορών που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον. Οι νέες μορφές κινητικότητας που βασίζονται σε οικονομικά συνεργατικής οικονομίας επίσης θα πρέπει να προωθηθούν. Θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε η φορολόγηση της ε, χρήσης ε, των ποδηλάτων ε, και της χρήσης των δημοσίων μεταφορών. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν περιοχές όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις, οπότε δεν θα πρέπει να τιμωρούνται και οι αυτοκινητιστές. Θα πρέπει να αποφύγουμε διακριτική μεταχείριση κατά οποιοδήποτε τρόπο μεταφοράς και κυρίως να σεβόμαστε την αρχή της επικουρικότητας, διότι θεωρώ ότι η εφαρμογή της πολιτικής κινητικότητας ε, είναι αρμοδιότητα των Δήμων και κοινοτήτων. Δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε ομοιόμορφη λύση. Έληξε ο χρόνος σας, κύριε μου, κύριος Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι επίγον να αντιμετωπίσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές και στα πλαίσια της COP21 η Ευρώπη πρέπει να είναι πρωταγωνιστή στο Παρίσι αλλά δυστυχώς οι παραγωγοί δεν βοηθούν. Μετά το σκάνδαλο Volkswagen, από ό,τι φαίνεται το ποσοστό δείκτη συμβατότητας αυτό το 2,1 δεν είναι αντίστοιχο με τους κινητήρες Euro 6 ε, και εξακολουθούν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα και να παράγονται πόσο μάλλον αυτοκίνητα τα οποία έχουν υπερδιπλάσιες ε, εκπομπές ε, ε, διαφόρων διοξιδίων όπως λοιπόν λέγει και η συγγήτρια νομίζω ότι το θέμα της αηφορίας στην κινητικότητα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την αντιμετώπιση των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Κύριος Κέλλη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στα πλαίσια της COP21 ε, και χαίρομαι που θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η συζήτηση. Μιλάμε για την κυκλική οικονομία και τώρα περνάμε και στην αισθητική κινητικότητα σχετικά αλληλένδετα ζητήματα. Φυσικά αυξάνεται το ποσοστό των αριθμών που το ποσοστό των πολιτών που ζουν σε τέτοιε περιοχέ οπότε είναι ιδιαίτερα επίκαιρο το ζήτημα και φυσικά θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτησή μα από τα ορεκτά καύσιμα και ε, να απομακρυνθούμε από τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στο μέτρο του δυνατού. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στις ε, κομίτείε που γνωρίζω εγώ στη χώρα μου. Έχουν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες, ε, όχι μόνο για τι μεταφορέ, αλλά και για την ανακύκλωση και γενικότερα με δράσει φιλικέ προ το περιβάλλον. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν. Υπάρχουν ε, μεταφορέ που πρέπει να γίνουν μέσω των πολλών και αυτό που πρέπει να φροντίσουμε είναι να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα ζωή και να επιστρέψουμε τι πόλει στου πόλει. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα σχέδια βιώσιμη αστική κινητικότητα είναι άμεσα συνυφασμένα με την προώθηση τη βιώσιμη αστική συγκοινωνία δεδομένου ότι σύντομα το 80% των ευρωπαίων θα ζουν σε πόλεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 30% των σοβαρών τραυματισμών από τροχαία λαμβάνει χώρα σε αστικές περιοχές θα πρέπει αρχικά να εξασφαλιστεί τόσο η προσβασιμότητα στην εργασία και στις υπηρεσίες για όλους όσο και η ασφάλεια στην κινητικότητα των πολιτών. επιπλέον θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η οικονομική αποδοτικότητα των μεταφορικών μέσων και να αυξηθεί η ελκυστικότητα του αστικού περιβάλλοντος γενικά. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει κάθε τοπική αρχή και να αυξήσει τη χρηματοδότηση της αστικής κινητικότητας ώστε να βελτιωθεί. Καθώς το 40% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα οφείλεται σε κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται στις μεγάλες πόλεις, θα πρέπει να οριστούν δεσμευτικοί στόχοι που να αφορούν τη μείωση των ρήπων που προκαλούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας ε, την εισηγήτρια και όλους τους κοιόδους εισηγητές. Ε, πιστεύω πως το κλειδί της λύσης για μακροπρόθεσμα προβλήματα, τα προβλήματα εκπομπών συγκεκριμένα στις πόλεις, έχουν σχέση με την καλύτερη οργάνωση των αστικών μεταφορών και περιαστικών μεταφορών. Οι καλές δημόσιες μεταφορές μπορούν να καλύψουν και την αυξανόμενη ζήτηση με καλύτερο σχεδιασμό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τις ε, νέες τεχνολογικές εξελίξεις και την τηλεματική. Ε, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ευάλ... τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που εξαρτώνται από τις δημόσιες μεταφορές. Χρειαζόμαστε κατάλληλη υποδομή για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, στην Κροατία ε, πριν από 15 χρόνια εγώ οργάνωσα την πρώτη ημέρα χωρίς αυτοκίνητα. Ε, επιτύχαμε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια να αυξήσουμε τη χρήση των δημοσίων μεταφορών. Αυτό έχει συμβεί και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ε, όμως, δυστυχώς, στον τομέα τη αστική κινητικότητα αυξάνονται διαρκώ ε, οι εκπομπέ των αερίων του θερμοκηπίου και ε, τέσσερις στους πέντε πολίτες ε, σύντομα θα μένουν ε, σε αστικά περιβάλλοντα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωή και το περιβάλλον. Σε πολλέ περιοχέ συνεχίζουν να έχουν την πρωτοκαθεδρία τα αυτοκίνητα. Υπάρχει μεγάλη χορύπανση και αυξανόμενο αριθμό ατυχημάτων. Χρειαζόμαστε επανασχεδιασμό τη πολιτική αστική κινητικότητα και των δημοσίων μεταφορών για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να βασιζόμαστε σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ούτω ώστε να έχουμε χαμηλότερε εκπομπέ. Οι μεταφορέ θα πρέπει να καθολικά προσβάσουμε. Σας ευχαριστούμε. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, βρίσκω ιδιαίτερα ικανοποιητική την έκθεση για την αστική κινητικότητα. Περιγράφει τις σημαντικότερες προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη και οι διαφορετικές περιφερειακές ανάγκες και να τονιστούν στην έκθεση. Όχι άνωθεν, αλλά να ερωτηθούν πρώτα οι υπεύθυνοι επιτόπου για την ανάπτυξη των διαφόρων ε, προσεγγίσεων. Αυτό θα βοηθήσει πολύ. Επίσης, στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προσφέρουμε και βραχυπρόθεσμες, ε, βραχυπρόθεσμες λύσεις, έτσι ώστε όσοι προσφέρουν και όσοι χρησιμοποιούν τις υποδομές και τις υπηρεσίες κινητικότητας να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα αυτά να είναι προστατευμένα. Ελπίζω η παρούσα έκθεση να θεωρηθεί ως αφορμή για περισσότερα, η χορήγηση περισσότερων κινήτρων για την ηλεκτροκίνηση και ιδίω για ηλεκτρικά λεωφορεία για τις ε, Σούλινγκ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό τα αστικά κέντρα να μπορέσουν να αναπτύξουν βιώσιμη κινητικότητα το δυνατόν συντομότερο. Έχουμε εκεί και σημαντικές καινοτομίες. Η βιώσιμη κινητικότητα στα αστικά κέντρα είναι η καλύτερη χρήση των διαφόρων τρόπων μεταφορών όπου ρόλο παίζουν και το ποδήλατο και το βάδισμα και οι δημόσιες μεταφορές και όλα αυτά. Όλα βεβαίως έχουν και πλονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ολλανδοί εμπειρογνώμονες έχουν καταδείξει ότι η βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι και ανέφικτη πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε η βιώσιμη κινητικότητα να μην εξισώνεται με εντατική άσκηση. Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί οι άνθρωποι λαμβάνουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Έχει έρθει η ώρα νομίζω να εξασφαλίσουμε πιο αποτελεσματικές πολιτικές και αυτές να ενταχθούν στην βιώσιμη κινητικότητα. Ο κύριος ε, Κρέμερ το αυτοκίνητο δολοφονεί τις πόλεις μας. Το 1972 ο νεαρός τότε δήμαρχος μονάχου Χαντιόχεν φόγκελ είχε πει ότι τα αυτοκίνητα καταστρέφουν τις πόλεις. Ακόμα και αν όλα τα αυτοκίνητα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά, ακόμα και αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτά λαμβάνουν τον ηλεκτρισμό από ανανεώσιμες ενέργειες, πάλι θα καταστρέφουν τις ε, πόλεις. 100 εκτάρια την ημέρα καταλαμβάνονται στη Γερμανία από δρόμους και άλλες υποδομές. Στις 8 Οκτωβρίου, 28 Υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και ομόφωνα μάλιστα τον οδικό χάρτη για τα ποδήλατα. Και ο ίδιος ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Υπουργός και ένα μέρος των φορτίων να μεταφέρεται με ποδήλατα. Φανταστείτε στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις να εξαφανιστούν τα μισά από τα φορτηγά. Τι ωραίο όραμα. Κυρία ε, Επίτροπε, τι μπορείτε να πράξετε για να δώσετε κίνητρα σε αυτά τα λεγόμενα cargo bikes, δηλαδή στα, ποδήλατα φορτίου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κύριο Σούγκαρ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. 23% των διοξιδίων, των διαφόρων καυσαερίων δηλαδή, προέρχονται από την κυκλοφορία των αστικών κέντρων και τα πράγματα επιδεινώνονται. Νομίζω ότι όλοι και όλες συμφωνούμε ότι η ανάπτυξη της αστικής κινητικότητας πρέπει να, είναι, να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και μέσα στην προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος και να ευθυγραμμιστούν να ευθυγραμμιστεί μάλλον η κινητικότητα με τις ανάγκες αυτές. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη πρέπει να προωθήσουν δοκιμασμένες πρακτικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Να θεσπίσουν μάλιστα και συστήματα δημοσίων προμηθειών που να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του περιβάλλοντος σε μεγαλύτερο βαθμό. Θα σε ευχαριστώ πολύ. Λίγη εδώ το λεγόμενο Catch Επανερχόμεθα σε εσάς κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους για τα σχόλια και τις παρεμβάσεις σας, καθώς και για ορισμένες ερωτήσεις που θέσατε. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω κάπως περισσότερο και να σας δώσω και ορισμένες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα που προτιθέμεθα να κάνουμε καθίσταται σαφές ότι είναι πολυδιάστατες οι προκλήσεις της ε, αστικής κινητικότητας. Το 2011 με τη Λευκή Βίβλο τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τον στόχο ανταγωνιστικής αστικής κινητικότητας. Το δε πακέτο του 2013 προσέφερε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίτευξη του στόχου. Με τη δική σας έκθεση όμως λαμβάνουμε νέα όθηση για την εφαρμογή του πακέτου αυτού. Με την υποστήριξή σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στους τομείς όπου η ευρωπαϊκή δράση μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία, βεβαίως με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Ιδίως σχεδιάζουμε να προωθήσουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση για ε, ευφυείς πόλεις και για ε, την προώθηση λύσεων καινοτόμων έργων για πραγματικές, ε, δηλαδή για δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες ε, λύσεων για τον ορίζοντα 2020 και να προωθήσουμε και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, για παράδειγμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αναφερθήκατε και εσείς σε φόρουμ για την ανταλλαγή πρακτικών στο ευρωπαϊκό επίπεδο που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Επιτρέψτε μου τώρα να απαντήσω σε ορισμένες από τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, για το φορτίο, για τα φορτία. Έχετε πλήρη υποστήριξη από μέρους μου. Το, η Λευκή Βίβλος του 2011 μιλεί για εφοδιαστική μηδενικών καυσαερίων ε, μέχρι το 2020 ή 2030 μάλλον. Άρα λοιπόν αυτά τα έχουμε υπόψη μας. Το δεύτερο ήταν για την τροχαία ασφάλεια. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ιδίως για τους πλέον ευάλωτους στον, ε, μέσα, μέσα στην τροχιά κυκλοφορία. Ήδη έχουν γίνει πολλά πράγματα, αλλά καθημερινά εμείς πιέζουμε τις χώρες μέλη να πράξουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με εκείνους που δείχνουν οι στατιστικές ότι βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση και συνεργαζόμαστε και με όλους τους ενδιαφερομένους στις διάφορες αυτές χώρες για να μειωθούν οι αριθμοί των θυμάτων όσο το δυνατόν να προσεγγίσουν δηλαδή το μηδέν. ποδήλατα. Όπως είπε ο κύριος Κράμερ αλλά και ορισμένοι άλλοι από εσά. Είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία των λύσεων πράσινη μεταφοράς φορτίων στις ε, πόλεις. Εμείς εξετάζουμε ε, ενδεχομένε επιλογές για να βελτιώσουμε την χρήση τους. Υπήρξαν και ορισμένα σχόλια ή ερωτήσει σχετικά με το καύσιμο δίζελ. Βέβαια πρέπει να βελτιωθεί το σύστημα διάθεσης στην αγορά των αυτοκινήτων, επίσης των εγκρίσεων τύπου. Χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί ελέγχου και των δοκιμών των αυτοκινήτων. Χρειάζεται να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή να ξεφύγουμε από τις δοκιμές εργαστηρίων και να προχωρήσουμε σε συνθήκες πραγματικές. Πιστεύω ότι θα συμβάλλει πολύ σε αυτή την προσπάθεια και η ηλεκτροκίνηση των ε, ε, αστικών μεταφορών. Σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πολυτροπικότητα με σωστό μείγμα, μια δηλαδή εκστρατεία για σωστό μείγμα, όπου περιλαμβάνει και το βάδισμα και, τα, και, την κίνηση με ποδήλατα και με δημόσια μέσα συγκοινωνίας και ούτω καθεξής. Κάτι που θα ωφελήσει όλες και όλους μας. Επιτρέψτε μου επίσης να επανέλθω σύντομα στα σχόλιά σας για την ποδηλασία. Ας μην υποτιμήσουμε τα οικονομικά ωφέλη από την ποδηλασία και για την υγεία και για την μείωση των καυσαερίων αλλά και βεβαίως και για την βιομηχανία. Καλωσορίζω λοιπόν την δήλωση του Συμβουλίου και εμείς σίγουρα θα κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή μέσα στα πλαίσια της εντολής μας. Ολοκληρώνοντας επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια ακόμη σχετικά ε, με το, σύστημα. Βεβαίως πρέπει να συνεργαστούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης έτσι ώστε να αλληλοσυνδεθούν καλά οι πόλεις και να γίνουν πράσινες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα στηρίξει την, ε, τις νέες ιδέες που αναφύονται. Βέβαια, τα ενδιαφερόμενα μέρη, stakeholder δηλαδή, μπορούν να προσφέρουν και νέες θέσει απασχόληση. Σα ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την υποβολή τη εκθέσεώ σα. Το 2016 Το δικό μου χαρτοφυλάκιο είναι το έτος της μείωσης των διοξιδίων του άνθρακος. Είμαι βεβαία ότι μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, της πρωτοβουλίας αυτής, θα περιλάβουμε και την ε, βιώσιμη κινητική ε, συγγνώμη, την βιώσιμη αστική κινητικότητα, για να βελτιώσουμε και τι συνθήκε διαβίωση στον πλανήτη μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ολοκληρώσει η κυρία Καριμά Να μου επιτρέψετε να σχολιάσω κάποια πράγματα τα οποία είπε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στην έκθεση δεν λέγεται απαγόρευση των αυτοκινήτων. Λέγεται απαγόρευση των αυτοκινήτων στα κέντρα των πόλεων, ιδιαίτερα αυτών με συμβατικά καύσιμα. Όπως ακριβώς το έλεγε και η λευκή Βίβλο στην οποία προώθησε ο κ. Βαντενκάμπ. Μη μας βάζετε λοιπόν λόγια ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι λύσεις οι οποίες προτείνονται στην έκθεση αυτή είναι ουσιαστικές, είναι πραγματικές. Ας προωθήσουμε στόχους συγκεκριμένους μέχρι το 25 για τα ποδήλατα. Ας αυξήσουμε τις ε, μαζικές μορφές συγκοινωνίας. Ας ε, προσπαθήσουμε να γενικεύσουμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητα Ας περιορίσουμε με πολύ φιλόδοξο τρόπο τα όρια ταχύτητας. Ας καταστήσουμε συμβατά τα ποδήλατα με τα αυτοκίνητα. Ας επενδύσουμε στην αστική κινητικότητα ε, ένα μεγάλο κομμάτι και του προγράμματος Juncker και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών ταμείων ας προσχωρήσουμε στη χρήση νέων ε, πρακτικών όπως ε, η αποκοινού χρήση ενός αυτοκινήτου. Ε, ας προβλέψουμε βελτίωση της νομοθεσίας για την ποιότητα του αέρα που αναπτέουμε. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που διώκονται φυσικά για τον μη σεβασμό των ανωτάτων ορίων και τα θύματα είναι οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι που είναι και θύματα των απατών των αυτοκινήτων βιομηχανιών σε σχέση με τη χρήση των πετρελαιοκινητήρων. Ας υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο σεβασμό στην υγεία των πολιτών και στην υγεία του πλανήτη. Σας ευχαριστώ κυρία Αντελή. Ε, διακόπτουμε για τρία λεπτά. Στις 7 ακριβώς θα ξεκινήσουμε.